έχει προβεί στην ε, επαλήθευση και επικύρωση ε, των εντολών του κύριου Παντάρ, κύριου Μόντου, κύριου Μάντλ και τέτοιων ε, σε συνέχεια της εντολής τους από 6 11, 8 11 και 30 11 17 και 1 πρώτου 18 αντιστοίχως. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις οπότε επικυρώνονται οι εντολές των συναδέλφων.